Ε, πρόκειται για ε, μια επίθεση στην ελευθερία τύπου που επίσης είναι μια αξία θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας και αυτό έγινε λίγους μήνες μόλις μετά την δολοφονία της Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια της Μαλτέζας δημοσιογράφου. Ο Κρούσακ με θάρρος ασκούσε το λειτουργήμά του και κατά την ε, διάρκεια αυτής της πολλαποσχόμενης καριέρας ασχολήθηκε με φοροδιαφυγή και φερόμενες υπεξαιρέσεις και δεν υποχωρούσε μπροστά σε τίποτα η αστυνομία δήλωσε ότι είναι βέβαιο το ότι δολοφονήθηκε για να σταματήσει τις έρευνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι όλοι θα πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα του για την ε, αλήθεια. Είναι απαράδεκτο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δολοφονείται δημοσιογράφος διότι επιτελεί το λειτουργήμά του. Και πρέπει να καταδικάσουμε όποιους εκφοβίζουν, φυλακίζουν τους ε, δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο. Ε, κατά τον εγγύσεων για ελευθερία του τύπου και κατά του ότι θα πρέπει με ασφάλεια οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι να ασκούν το επάγγελμά του. Και οι Σλοβακές Αρχές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια ε, και με τη βοήθεια διεθνούς συνεργασίας, ε, με συνεργασία με άλλες αστυνομίες. Και ακριβώ όπω και με την Δάφνη Καροναγκαλίτσια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα σταματήσει να διατρανώνει το ότι θα πρέπει οι ένοχοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και ακριβώς όπως ε, και με την περίπτωση της Μαλτέζας δημοσιογράφου θα πρέπει να τηρήσουμε ενός λεπτού υγεία. Grazie. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Purtroppo l'ultima settimana è stata densa di notizie. Δυστυχώς την προηγουμένη εβδομάδα είχαμε πάρα πολλά κακά μαντάτα. Οι Μπόκο Χαράμ, οι τρομοκράτες και πάλι επιτέθηκαν σε ένα σχολείο στην βορειοανατολική Νιγηρία και ε, πάνω από 100 ήταν τα θύματα, πάντοτε μιλάμε για παιδιά και οπότε και δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε αυτούς που το 2014 πήχθησαν από το τσίμπο γίνες οι κοπέλες. Εμείς καταδικάζουμε αυτή την επίθεση και επίσης επευθύνουμε έκκληση για την ε, απελευθέρωση των ε, ομήρων. Θα πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο. Με ασφάλεια και ελευθερία. Ο πρόεδρος ε, Μποχάρη είπε ότι πρόκειται για εθνική τραγωδία. Αλλά θα πρέπει εμείς να πούμε ότι πρόκειται για παγκόσμιο χαρακτήρα ανθρωπιστική τραγωδία. Επομένω θα πρέπει να δεσμευτούμε ακόμα περισσότερο πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά μαζί με τους ε, Αφρικανούς φίλους για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Σας ενημερώνω για ένα επεισόδιο που είχε πρωταγωνίσει πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλγαρία την συνάδελφο Σκακέλερ. Και είχαμε δήλωση του Υπουργού Σίμεροφ και επειδή συμμετέσχε σε κάποιο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά κάποιων εγκαταστάσεων στο Πυρήν ε, ζητήθηκε από την κυβέρνηση να απελαθεί. Ε, ήρθαμε σε επαφή με την κυβέρνηση και μας διαβίωσαν ότι αυτό δεν είναι θέση της κυβέρνησης και άρα δόθηκε λύση στο πρόβλημα. Είναι βασικό δικαίωμα η έκφραση της νόμης για οποιονδήποτε Ευρωπαίο και κυρίως για κάποιον που σαν την Κέλλερ ε, είναι ερετός, έχει εκλεγεί απευθείας από τους πολίτες, είναι αυτό για την ε, δημοκρατία μας. Κάποιος εκτός μικροφώνου ε, φωνάζει, οπότε μπορεί και να διαμαρτυρηθεί, είναι και αυτό δικαίωμα. Και ευχαριστούμε για την βουλγαρική κυβέρνηση που κράτησε αποστάσεις από αυτό το επεισόδιο και ευχόμαστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον. τι, τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ιδιαίτερος ε, τα σχόλιά σας. Λυπάμαι όμως που αυτή η ελευθερία έκφρασης δεν γίνεται σεβαστή και εντός του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και λυπούμε ιδιαίτερος που η νομική επιτροπή που εξετάζει τα θέματα αυτά έρει συστηματικά αρσιασιλίας ε, βουλευτές του, ε, της μειοψηφίας μας όταν έχουν διαφορετική γνώμη από την πλειοψηφία. Δεν συνέβαινε αυτό όταν πρώτον μπήκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τότε ήταν ο κανόνας η έκφραση πολιτικής γνώμης να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δίωξη. Ε, πολλό δε μάλλον όταν γινόταν από έναν ε, ευρωβουλευτή για τους πολιτικούς αντιπάλους του. Τώρα έχουμε τελείως διαφορετική κατάσταση. Ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές υφίστανται κυρώσεις όχι επειδή διαταράσσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά λόγω των δηλώσεων που έκαναν. Όσο α, αμφισβητούμενες και αν είναι, όσο αμφιλεγόμενες και αν είναι, κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην ίδια την πεμπτουσία του κοινοβουλευτικού βίου, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί μας αναφέρεται εδώ το επεισόδιο με τις κοπέλες και την Μπόκο Χαράμ θα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά της ε, εκπαίδευσης έχουμε δεσμευτεί για να καταπολεμήσουμε την Μπόκο Χαράμ να κάνουμε κάτι για την απαγωγή για αυτές τις κοπέλες οπότε θα πρέπει να δούμε Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι με την παιδεία. Θα ε, ακουστεί η άποψή σας όταν έρθει η ώρα. Ήδη έχουμε και τη συζήτηση για το Πορετές πλαίσιμο και θα συζητήσουμε και για την Αφρική. Κύριε Χριστοφόρο. Αυτό το βήμα, το ισχυρό βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράζει τη βούληση και τη θέληση όλων των λαών τη Ευρώπη από το Ευρωκοινοβούλιο που είναι ο θεματοφύλακα και ο προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεσμών, αρχών και αξιών, να καταγγείλω. Μια χώρα η οποία θέλει να γίνει και χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαρκώ παραβιάζει κάθε αρχή κανόνα δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέσει και αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια τη χώρα τη που εισβάλλει στο Αφρίν που κατέχει εδώ και 43 χρόνια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αυτές τις μέρες εισέβαλε παράνομα, πειρατικά και τρομοκρατικά στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, παρεμποδίζοντας τις έρευνες για ανέβρεση φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και στη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη, παρεμποδίζοντας Ιταλικών συμφερόντων της εταιρείας ΕΝΗ, το ΣΑΙΠΕΜ 12.000, να προχωρήσει στη διερεύνηση των ενεργειακών πόρων στο οικόπεδο 3 το οποίο είναι αδειοδοτημένο. Χρησιμοποίησε πολεμικό στόλο και με πειρατικό τρόπο έξι πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Μπλόκαραν και παρεμπόδεσαν την έννοια στο να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της και την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω καταρχήν τις απεριόριστες ευχαριστίες του κυπριακού λαού για την άμεση παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσά προ καταδίκη τη Τουρκία. Όμω εδώ, σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να πούμε στην Τουρκία ω εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πλήττει τα συμφέροντα όχι μόνο μια χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα συμφέροντα τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ενεργειακά αποθέματα είναι αποθέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλει να τα υπερασπιστεί. Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι η Total και η Ένη Ευρωπαϊκών Συμφερόντων και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα περασπιστεί Και η Τουρκία δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα από τη γλώσσα των κυρώσεων. Και οφείλουμε εμεί όλοι εδώ να πούμε στην Τουρκία ότι με τέτοιε πειρατικέ ενέργειε δεν μπορεί να ζητά αναβάθμιση τελωνιακή ένωση, δεν μπορεί να ζητά το visa liberalization και δεν μπορεί να έχει μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Il Ανέκαθεν ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου για την εξαρτησία της Κύπρου και για τον σεβασμό του ε, δικαιώματος αλλά επίσης και για κάποια υποψήφια χώρα όπως η Τουρκία γιατί έχουμε επανειλημμένη τη επαφή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Και τώρα ε, αρχίζει... Α, πρώτα κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεδομένης κατάσταση στη Βενεζουέλα, περίπου 8.000 ε, πολίτε Ευρωπαϊκή ε, Καταγωγή ε, βρέθηκαν στη Μαδέρα, που είναι εξόχω απόκεντρη περιοχή τη Ευρώπη. Μια και είναι εδώ ο Επίτροπο, ε, θα ήθελα να πω τι μέτρα πρόκειται να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει αυτή την τόσο μικρή εξόχως απόκεντρη περιοχή που υποδέχεται όμως τόσο μεγάλο αριθμό ε, μεταναστών. Ευχαριστώ. Vorremmo chiederlo alla Commissione europea che è impegnata una Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει μια στρατηγική για τη μετανάστευση και επίση κατά το επόμενο πολιτέ δημιουργικό πλαίσιο θα υπάρξει σχετική δέσμευση για να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό. Νόμιμη μετανάστευση, παρόν μετανάστευση και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη μετανάστευση από την Αφρική. Συνεχίζεται τώρα η σύνοδος, η οποία 8 Δευτέρου είχε διακοπεί και έχουμε